Εγώ είμαι διατεθειμένη να το κάνω αυτό. Ε, θα ήθελα να ακούσω και από εσά αν είσαστε κι εσεί διατεθειμένοι να κάνετε το ίδιο και πώς, ε, ποια είναι η θέση σα για το θέμα της υπερβολικής ελευτική ικανότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φράγα. Sí. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Οι προηγούμενες ε, μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ σε μεγάλο βαθμό ναυάγησαν και απέτυχαν γιατί ποτέ δεν τροποποίησαν το τρόπο διαχείρισης των αλληλευτικών πόρων. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί διαφορετική θέση και πιστεύω ότι η νέα της θέση είναι αρκετά λογική. Κατά τη γνώμη μου αυτό το σύστημα είναι το μοναδικό σύστημα που μέχρι στιγμής ε, έχει δείξει καλά σημεία λειτουργίας. Και έχουμε πρόβλημα υπερβολικής ε, ε, ελευτικής ικανότητας που οδηγεί σε υπεραλίευση και άρα σε μη αηφόρο διαχείριση των ελευτικών πόρων. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Υπεραλίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω ε, ορισμένοι παρόλο που αναγνωρίζουν τα προβλήματα δεν θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση. Ενώ αυτό το σύστημα είναι το μόνο που είναι ικανό να αντιμετωπίσει τι νέε προκλήσει. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα διαχείριση. Ε, απέτυχε το μέχρι τώρα σύστημα διαχείριση. Αν δεν είχαμε υπερβολική ελευτική ικανότητα, δεν θα είχαμε υπεραλίευση. Αλλά υπάρχει και υπερβολική ελευτική ικανότητα και πλεονάζουσα ικανότητα και υπεραλίευση. Όλοι το διαπιστώνουμε στα σε 99,9% των περιπτώσεων δεν είχαμε ε, λιγότερη ε, αλληλευτική ικανότητα. Ο κανόνας είναι πλεονάζον δυναμικό, πλεονάζον αλληλευτική ικανότητα και μην μου λέτε ότι δεν ισχύει αυτό. Κάποιος θα πρέπει να επινοήσει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης. Το μοναδικό μοντέλο διαχείρισης που μας επιτρέπει πραγματική μείωση της αλληλευτικής ικανότητας είναι το μοντέλο αυτό τον. Ε, ε, TFC που προσαρμόζεται στις διάφορες συνθήκες. Αν λοιπόν στόχος μας είναι η μείωση της υπεραλίευσης και του πλεονάζοντος δυναμικού στην αλία, το μοναδικό σύστημα που έχει δείξει κάποια στοιχεία αποτελεσματικότητας είναι αυτό. Εντάξει, μερικοί μίλησαν για συγκέντρωση κτλ. Αλλά για αυτό το ζήτημα, για να αποφύγουμε τη συγκέντρωση, έχουμε τις ρήτρες διαφύλαξης, διασφάλισης, για να αποφύγουμε τέτοια συγκέντρωση. Είμαι υπέρ των ρητρών για να αποφύγουμε τα προβλήματα συγκέντρωση, ακόμη και εντό του ίδιου κράτου μέρου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τι ρήτρε. Οτιδήποτε το δέχομαι, γιατί θεωρώ ότι το σύστημα αυτό είναι αποτελεσματικό. Και φυσικά θα το ελαστικοποιήσουμε. Κανένα σύστημα δεν λειτουργεί άψογα από την αρχή. Προσαρμόζεται σταδιακά στι νέε συνθήκε και στην πραγματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα θα λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα σε κοινοτικό επίπεδο. Αλλά ακόμη και τη ρήτρα για εθνική λειτουργία θα μπορούσα να τη δεχτώ. Αλλά είναι το καλύτερο μοντέλο μέχρι στιγμή. Οι τελευταίε μα εμπειρίε δείχνουν ότι οι χώρε που έχουν περισσο... του περισσότερου στόχου ε, προστασία περιβάλλοντο ε, και φόρου αελία, όπω είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ισλανδία, Καναδά, ε, Δανία, εφαρμόζουν αυτό το σύστημα και μάλιστα με πολύ θετικά αποτελέσματα. Στην Νορβηγία είχαμε μείωση ε, κατά 50% του στόλου ε, ανοιχτή θάλασσα και 38% ε, της υπεράκτης ελίσμας στους 5 ε, ε, χρόνια. Τα ποσοστά ρέγγας μειώθηκαν κατά 50% σε 4 χρόνια. Στην Ισπανική, στον Ισπανικό ε, λευτικό στόλο, όταν εφαρμόστηκε σε ένα είδο και πάλι είχαμε μείωση κατά 50%. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, έχουμε οδηγηθεί σε μείωση τη αλληλευτική ικανότητα. <clears throat> Άλλωστε, αυτό δεν γίνεται με κανονιστικό τρόπο. Αυτή η μείωση της ε, αλληλευτικής ικανότητας γίνεται με επιχείρημα... απόφαση της επιχείρησης. <clears throat> Το κοινωνικό ζήτημα τώρα. Όντως μπορεί να έχουμε και κοινωνικές συνέπειες. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ χειρότερα τα κοινωνικά αποτελέσματα αν διονύσουμε το ισχύον σύστημα. Γιατί εκεί είναι που θα αποδεκατήσουμε τον αλληλευτικό μας κλάδο. Τώρα, όσοι είναι υπέρ του στάτου κβο μιλούν για τις επιδοτήσεις. Ε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το ισχύον σύστημα, αποκλείεται να επιβιώσουν χωρί επιδοτήσει οι αλληλεί. Οπότε θα χρειαστεί να, να διατηρήσουμε και τι επιδοτήσει. Τώρα υπάρχουν προβλήματα παγκοσμίω με τη διατήρηση των επιδοτήσεων. Τι έδειξε το ισχυρό σύστημα επιδοτήσεων και αυτό αναποτελεσματικό είναι γιατί δόθηκαν τεράστια κονδύλια αλλά δεν οδηγηθήκαμε στην επιθυμητή μείωση του αλληλευτικού δυναμικού. Κυρία Ρόντου, συμφωνώ απόλυτα με το νέο σύστημα. Και όποιο πρόβλημα έχουν οι συνάδελφοι, να το λύνουμε με τι ρήτρε διασφάλιση. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δεχτούμε αυτή την αρχή και μετά να θεσπίσουμε ρήτρε για να αποσοβηθούν οι φόβοι και οι ανησυχίε. Είμαι υπέρ τη αρχή. Βάλτε όσε ρήτρε διασφάλιση θέλετε. Ε, Ευχαριστώ κύριο Ντέιβιτ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτω και με την κυρία Ρόντοστ και με την κυρία Φράγα με ευχαριστεί ιδιαίτερα και με εκπλήσει το ότι σύμφωνο απολύτως. Μιλάμε για περιφερικοποίηση πάρα πολύ και λέμε ότι υπάρχει ανεπαρκής χρήση του όρου, αλλά εδώ έχουμε την καλύτερη ευκαιρία. Τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τους αλλιευτικούς τους στόλους και στα πλαίσια των εθνικών τους αλλιευτικών πολιτικών να θέτουν και κάποια κριτήρια οικονομικά και περιβαλλοντικά, παράλληλα με τα ευρωπαϊκά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε όλοι είναι ότι τα TFCs μπορούν να διαμορφωθούν και να ελεγχθούν. Δεν είναι ένα επιβαλόμενο εκ των άνω μοντέλο για όλες τις χώρες. Να απευθυνθώ περισσότερο στον κύριο Καντέκ γιατί ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι' αυτά. Έχω κάποιες τροπολογίες εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την επόμενη Τετάρτη θα τις καταθέσω κάποιες συγκεκριμένες ιδέες έτσι ώστε να κατευθύνουμε κάπως τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι το σημείο κίνησης μένει πάντα ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέσουν και να αποφασίσουν τους δικούς τους στόχους για τα TFC και για τις χρηστές πρακτικές τις οποίες θέλουν να συμπεριλάβουν σε αυτή. Κάνοντας τον σχεδιασμό των προγραμμάτων τους μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των ποσοστώσεων που μπορούν να διανεμηθούν και να αναδιανεμηθούν 10, 15, 20%. Μπορούν να προσαρμόσουν τα TFC σε συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή οι παράκτιοι δεν θα μπορούν να έχουν και πελαγικές άδειες κτλ. Επίσης μπορούν να ρυθμίσουν καλύτερα τις αιτήσιε ε, ποσοστώσεις. Πρέπει να είσαι ο ίδιος ε, Ε, ε, εμπλεκόμενο στον τομέα της αλίας. Δεν μπορεί να λέμε ότι η Manchester United σαν παράδειγμα υποτίθεται από ό,τι ακούγεται ελέγχει πάρα πολλές εκχωρήσεις και αδειοδοτήσεις στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορούμε ας πούμε να ε, δεσμεύουμε ένα μικρό τμήμα των TFCs για τους νέους που μπαίνουν στην αγορά κάθε χρόνο. Και μια ολόκληρη σειρά από άλλα νομικά μέτρα τα οποία μπορούν να εισάγουν έτσι ώστε να μην καταλήξουμε τελικά ε, με την απλή ιδιοκτησία των TFCs από φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με την αλληλεία. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά προστατευτικών μέτρων τα οποία θα πρέπει να εισάγουν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Τελικά ποια είναι η ουσία και το έθεσε πολύ καλά η κυρία Φράγα. Τα TFCs δουλεύουν, δουλεύουν και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Τα αλλιεύματα έτσι και αλλιώ ανακάμπτουν και στην Ισλανδία και την Νορβηγία και ο κόσμος που δεν του αρέσει το TFC πρέπει να μας δώσει εναλλακτικές προτάσεις. Κύριο Καντέκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα εκπλαγείτε ότι εγώ δεν συμφωνώ ούτε με την κυρία Φράγα, ούτε με, με την κυρία Ρόντουστ, ούτε με τον κύριο σχετικά με τις ε, μετατίευσεις, τις μεταφερόμενες αδειοδοτήσεις. Αυτές οι αδειοδοτήσεις εφαρμόζονται σε όλα τα αλλιευτικά σκάφη άνω των 12 ε, μέτρων, μέτρων και επίσης ε, και σε κάτω από 12 μέτρα εφόσον είναι εξοπλισμένα με συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, δηλαδή όλα τα αλλιευτικά σκάφη. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον έχουμε πάντα σαν στόχο τη διατήρηση των αλλιευμάτων, αυτό θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαχείρισης από τις οργανώσεις των παραγωγών ή τις δημόσιες αρχές. Όχι σε νομισματική βάση όταν υπάρχουν αλλαγές, να μην γίνονται οι αλλαγές αυτές σε νομισματική βάση. Το νομισματικοποιημένο μεταφερόμενο σύστημα διοδοτήσεων σας έχω πει ότι είναι κακή επιλογή. Εγώ επαναλαμβάνομαι, αλλά η νομισματικοποίηση των φυσικών πόρων, η υπερβολική συγκέντρωση των δικαιωμάτων στις μεγάλες εταιρείες και μεσοπρόθεσμα, είτε το θέλουμε είτε όχι, στην εξαφάνιση της παράκτιας αλληλείας η οποία παίζει πάρα πολύ ε, σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση της υπαίθρου σε παράκτιες περιοχές. Αναφερθήκατε στην Ισλανδία, Ξέρετε τι συμβαίνει εκεί δυστυχώς. Επίσης παράλληλα θα υπάρξει και μια κερδοσκοπική χρήση των αδειών, μια πλήρης απορρίθμιση και απελευθέρωση και μια αγορά νέα ε, ανταλλαγής δικαιωμάτων ανάμεσα σε χώρες. Κοιτάξτε, στόχος μας είναι ε, πάντα η διατήρηση των αλλιευμάτων και όχι η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων που θα επιφέρει περιβαλλοντική και οικονομική χειροτέρευση. Δεν θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν το σύστημα που θα αποφασίζουν. Κάθε κράτος μέλος θα αποφασίζει στο δικό του εθνικό πλαίσιο. Μιλήσατε για την περιφερικοποίηση. Εγώ δεν το προτείνω αυτό. Δεν μπορούμε να εργαστούμε μόνο σε περιφερειακό επίπεδο. Πάντως συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπευθυνοποιηθούν οι αλληλείς, σαφώς, αλλά εκτός της νομισματικοποίησης εισαγωγικά των δικαιωμάτων. Σχετικά με τις μεταφορές, θυμίζω ότι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 επιτρέπεται η μεταφορά διοδοτήσεων ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Ενώ στο παρελθόν, αν ενθυμίστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε πει ότι θα πάρει μέτρα για να μην συγκεντρωθούν τα δικαιώματα σε ορισμένες χώρες, κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει. Γνωρίζετε τις γνώμες μου λοιπόν για τα TFCs, είμαι κατά για τους λόγους που ανέφερα τώρα, που προανέφερα και στο παρελθόν και που θα αναφέρω και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Καντέκο. Κύριε Σφερέρα, ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, η θέση της κυρίας Ροντού ότι το είναι ότι το σύστημα θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Δηλαδή να εναπόκειται στα κράτη-μέλη αν επιθυμούν να το εφαρμόσουν. Αν κατάλαβα καλά, η θέση της ηγήτριας ε, είναι αυτή, προαιρετική εφαρμογή. Αυτό διαφέρει από τις θέσεις ε, των κυρίων Φράγκα και Ντέιβιτς, με τους οποίους διαφωνώ ριζικά. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε πλέον πρώτα μια περιστατευμένη γνώμη της κατάστασης πριν να προβούμε σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Για την υπερβάλλουσα αλληλευτική ικανότητα είπε ότι μειώνεται όταν ε, εφαρμόζεται το σύστημα μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων. Πού όμως, για, ε, για ποια τμήματα του αλληλευτικού στόχου δεν είναι ισχύει. Δεν νομίζω ότι είναι πλήρης εικόνα που έχουμε για τα διάφορα αυτά στοιχεία. Πρώτα θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να έχουμε πλήρη γνώση κατάσταση και μετά να εφαρμόσουμε ένα δίκαιο σύστημα. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε γενικούς ορισμούς και να λέμε γενικά και αόριστο ότι έχουμε υπερβάλλον ελευτικό δυναμικό. Πού, σε ποιες περιοχές, για ποιους ελευτικούς στόλους, για ποια ελευτικά είδη. Θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουμε όλα αυτά τα κενά που έχουμε στη γνώση. Και μετά, ε, αν όντω διαπιστώσουμε γενικευμένη αλληλευτική υπερβάρουσα αλληλευτική ικανότητα, τότε να δούμε τι μέθοδο θα εφαρμόσουμε. Υπάρχει μία μέθοδος ε, νομοθετική, κανονιστική και ίσως θα πρέπει οριζόντια να μειώσουμε το ελευτικό δυναμικό κατά χ% ας πούμε. Οπότε αυτή η κανονιστική μέθοδος θα πρέπει να αποφασίσει ποιες, ποιες θα αποκλειστούν. Υπάρχει όμως και η μέθοδος αγοράς που λέει η αγορά θα αποφασίσει ποιες, ε, που θα γίνουν οι περιορισμοί. Αναφέρθηκε το πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα και η σύγκριση που έγινε ε, με το σύστημα είτε των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων είτε με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Έγιναν παραλληλισμοί ε, αυτών των συστημάτων. Βέβαια, η συζήτηση έγινε σε νομικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικός αυτός ο παραλληλισμός. Για τα καυσαέρια, και εκεί έχουμε για το σύστημα εμπορία εκπομπών δύο ε, επιλογές. Έχουμε την κανονιστική ρύθμιση που μειώνει με νομοθεσία το ύψος των καυσαερίων και λέει στους φορείς ποιο είναι το ανώτατο όριο που επιτρέπεται να εκπέμπουν καυσαέρι και υπάρχει και η λύση της αγοράς. Η λύση της αγοράς είναι αυτή που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύστημα εμπορία εκπομπών. Βέβαια, οι συνέπειε είναι διαφορετικέ. Όπω είπε η κυρία Φράγκα, μα μίλησε για τι συνέπειε ε, τη προσέγγιση αγορά. Θα φύγουν ε, οι αναποτελεσματικοί αλληλεί, οι αναποτελεσματικοί στόλοι και θα επιβιώσουν οι πιο ικανοί. Αυτό που θα αποφασίσει η αγορά είναι να παραμείνουν οι πιο τα πιο αποτελεσματικά σκάφη, από αμυγή όμως οικονομική άποψη μόνο με βάση το οικονομικό κριτήριο θα επιβιώσουν κάποια ηλιευτικά σκάφη. Η όμως μας ορισμένες χώρες, όπως είπε ο κ. έδειξε ότι τα πλοία που παροπλίστηκαν ήταν αυτά που από περιβαλλοντική άποψη και από κοινωνική άποψη ε, είτε λόγω του χαμηλού αντίκτυπου, είτε λόγω του θέσης απασχόληση, ήταν αυτά που ενίσχυαν την αηφόρα αλία. Ε, Τελικά αυτά τα σκάφη που παρέμειναν ήταν τα πιο αποτελεσματικά από οικονομική άποψη, αλλά όχι τα πιο αποτελεσματικά από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Αυτό έδειξε η εμπειρία μας όταν αφήνουμε την αγορά να αποφασίζει, όπως γίνεται με ένα τέτοιο σύστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ρήτρες διασφάλισης, δεν υπάρχει ούτε μία ρήτρα διασφάλισης που να σταθμίζει τη ε, συνέπειση να αποσοβεί την ε, συγκέντρωση. Να περιορίσουμε τις άδειες σε συγκεκριμένο επιχειρηματία. Ναι, αλλά κάθε επιχειρηματής μπορεί να έχει πολλές και διάφορες επιχειρήσεις και κάθε επιχείρηση να αγοράζει ξεχωριστά τις παραχωρήσεις. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να, παραμε... να ε, ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Κανένας δεν εμποδίζει και άλλους ε, που μη λύση ε, εφοπλιστές, ε, που αχυρά άνθρωποι θα μπαίνουν στην αγοραπολισία αυτή και θα αγοράζουν τέτοιες μεταβιβάσεις ελευτικών παραχωρήσεων, τέτοιες άδειες ελευτικές. Ούτε και αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Επίσης, ο πάροχος ε, ενός, ε, ε, φορές ενός συγκεκριμένου μέλους, ένα επιχειρηματή συγκεκριμένου μέλους, κάλλιστα θα μπορούσε να πάει σε άλλο κράτος μέλος και να αγοράσει τέτοιες άδειε. Δεν μπορούμε όλους αυτούς τους κινδύνους να τους αποσοβήσουμε με ρήτρες διασφάλισης. Όποιες ρήτερε διασφάλισης και να εφαρμόσουμε, δεν, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη συγκέντρωση. Αποκλείεται. Υπάρχουν πολλά μέσα για να την καταφέρουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον παραλληλισμό με τι γαλακτοκομικέ ποσοστώσεις και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία Εκπομπών. Α δούμε τι συνέπειε και των δύο συστημάτων. Τι έγινε με τι γαλακτοκομικέ ποσοστώσεις. Μειώθηκε η γαλακτοπαραγωγή. Όχι, το αντίθετο αυξήθηκε. Είχαμε όμω συγκέντρωσή τη σε λίγου επιχειρηματίε. Στην Πορτογαλία 70-80.000 ε, παραγωγή γάλακτος ε, αποδεκατίστηκαν τα τελευταία χρόνια, εξαφανίστηκαν. Αντίθετα, η γαλακτοπαραγωγή δεν μειώθηκε, το αντίθετο. Τι γίνεται με τι άδειε τη ε, εμπορία εκπομπών. Είχαμε μείωση των καυσαερίων από το 2005 που εφαρμόσαμε το σύστημα. Όχι, αντίθετα, είχαμε αύξηση των καυσαερίων. Τίποτα λοιπόν δεν μας βεβαιώνει ότι το σύστημα αυτό των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων θα μειώσει την ε, αλληλευτική προσπάθεια. Απλώς θα γίνει συγκέντρωση ενώ θα εξαφανιστούν πολύ μικροί αλληλείς. Δεν ε, επιθυμούμε μια τέτοια συγκέντρωση. Γιατί τελικά αυτή η συγκέντρωση θα, συγκεντρω... θα έχει ω συνέπεια όχι κατά ανάγκη τη μείωση, μπορεί να έχουμε και την αύξηση τη ελληνική προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν χάσει τη δουλειά τους πολλοί αλλοί. Νομίζω ότι αυτός ο παραλληλισμός είναι πολύ χρήσιμος και θα πρέπει να μας κρούσει τον κόδωνα, τον κόδωνα του κινδύνου. Νομίζω ότι εναλλακτική λύση και εναλλακτική μέθοδος σωστή είναι η κανονιστική μέθοδος, η νομοθετική ή να περιορίσουμε τις ε, άδειες ε, ε, αλίες, να περιορίσουμε αυτές που θα δοθούν στην αγορά. Μπορούμε νομοθετικά να αποφασίσουμε ποιοι τομεί θα μειωθούν, σε ποιες ώρες, σε ποια ληφτικά είδη και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα, η κυρία Βιλβάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική. Καταρχήν, συμφωνώ με τον κύριο Φερέιρα και παραλαμβάνω το αίτημά μου που είχα υποβάλει και στην ε, Επίτροπο Δαμανάκη που όταν υπέβαλε την πρόταση για την αναθεώρηση το είχα ζητήσει. Θα ήθελα να έχουμε μία σαφή ε, ανάλυση της κατάστασης για να γνωρίζουμε πλήρως τι συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ένα χάρτη, μία απεικόνηση της κατάστασης για να δούμε τι έγινε σε κάθε χώρα και κάθε ελευτικό στόλο τα τελευταία πέντε χρόνια. Για να δούμε ποια ήταν τα αποτελεσματικά συστήματα, πώς λειτουργήσαν τα μέτρα και πού δεν λειτουργήσαν. Εγώ συμφωνώ με το σύστημα μεταβιβάσιμων αλευτικών παραχωρήσεων, TFC, αλλά πιστεύω ότι έτσι θα έχουμε μία μείωση του αλευτικού στόλου με τεράστιες όμως οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Και αυτές οι συνέπειες δεν μπορούμε να τις ε, αγνοούμε. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με άλλες πρωτοβουλίες. Ναι, ε, λέω στα TFC, να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες της αναδιάρθρωσης, να επιζητούμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αλλά να μην εθελοτυφλούμε απέναντι στις ε, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες και να βοηθήσουμε κάπως ή να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των ζωνών που εξαρτώνται από την αλληλεία. Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση αλληλευτικών παραχωρήσεων θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και ε, για τι επιδοτήσει για, για τον παροπλισμό των πλοίων. Σε προηγούμενες συζητήσεις είπαμε ότι θέλουμε να ορίσουμε την ε, παράκτεια και την ε, αλία μικρής κλίμακος. γιατί η αλία αυτή έχει συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και οι τοπικές κοινότητες εξαρτώνται σχεδόν πλήρως από τέτοιου είδους παράκτη αλία. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Αυτή λοιπόν η θέση μου από τις αρχές. Εγώ είμαι υπέρ του συστήματος των μετεβάσεων αλληλευτικών παραχωρήσεων, αλλά με εχέγγυα, με ρήτρες διασφάλισης. Συμφωνώ με την κυρία Φράγκα. Χρειαζόμαστε ρήτρε διασφάλισης και εχέγγυα για να έχει το σύστημα αυτό τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα. Κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την κυρία Ρόντουστου που έθεσε τόσο σαφώς το ερώτημα, να σκεφτούμε δηλαδή το θέμα της ε, υπερβολικής ε, αλληλευτικής ικανότητας ε, και όχι να επικεντρωθούμε τόσο πολύ στο θέμα των μεταβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων. Εγώ δεν παθιάζω πολύ με το θέμα αυτό των TFC, διότι γνωρίζω ότι μπορεί να σχεδιαστεί το σύστημα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ε, και ξέρω ότι στην Νορβηγία ε, έχει ε, εφαρμοστεί πολύ καλά το σύστημα όπου είναι με περιφερειακή βάση και στις Ηνωμένε Πολιτείε όπου είναι με κοινοτική βάση. Όλα αυτά όμως έχουν εφαρμοστεί προαιρετικά στις Ηνωμένε Πολιτείε έχει εισαχθεί αναλύευμα σε προαιρετική βάση και στην Νορβηγία οι βουλευτές μαζί με τα μέλη του ελευτικού τομέα έχουν εισάγει το σύστημα αυτό βαθμιαία. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πούνε στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο. Μπορούν όμως να το κάνουν. Και θα μπορούσε να είναι καλή η αρχή, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πόροι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσης για τους ε, αλληλείς μικρής κλίμακας ε, για να μπορέσουν ε, αυτοί να οργανωθούν και να δουν πώς μπορούν να λύσουν το θέμα της υπερβολικής αλληλευτικής κανότητας. Θα πρέπει να εξετάσουμε ένα αλίευμα πόσο η περιττή αλληλευτική ικανότητα έχουμε και ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ήταν χρήσιμο εάν κατά την κατανομή ε, αλλιευτικών δυνατοτήτων μπορεί να αφισβητηθεί η χρήση της λογικής των ιστορικών αλλιευμάτων. Μπορεί να κοιτάξει κανείς αναλύευμα, δηλαδή τι είδους τι αλλιευτική ικανότητα έχουμε και ποια είναι η επιθεμητή αλλιευτική ικανότητα και να δοθεί ε, πρόσβαση προτεραιότητα σε, σε αυτούς που αλλιεύουν με τον κοινωνικά και οικολογικά πιο βιώσιμο τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει. Αυτό μπορεί να δώσει κανείς περισσότερες μέρες στη θάλασσα σε όσους έχουν ε, ε, θελοντικά επιλέξει να έχουν κάμερα κλειστού κυκλώματος, CCTV ή επιλεκτικά εργαλεία ε, εργαλεία αλίευσης ε, ή σε αυτούς ε, που, έχουν, που δεν έχουν ιστορικό παράνομης αλληλείας σε αντίθεση με αυτούς που έχουν ιστορικό παράνομης αλληλείας μην ξεχνάμε ότι τα ε, ψάρια ανήκουν στην κοινότητα στο σύνολό τους ε, και είναι πολύ σημαντικό να ε, θυμόμαστε την αρχή αυτή. Δεν θέλουμε να δούμε τις εξελίξεις που είδαμε στην Ισλανδία όπου λίγο πολύ κάποιες ξένες τράπεζες είναι ιδιοκτήτες των αλλιευτικών πόρων και έχουν πρόβλημα για το, σχετικά με το πώς μπορούν να επανεθνικοποιήσουν τα ψάρια τρία πράγματα στο κείμενο της Επιτροπής. 15 χρόνια που προτείνονται, νομίζω ότι είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Δανία έχει 8, η Σουηδία έχει 10 για την ε, πελαγική αλληλεία. θα ήταν πρόβλημα για μας αν περάσει ε, αυτή η διάρκεια. Επίσης, όσον αφορά την, ε, το ανώτατο όριο της αλληλευτικής ικανότητας, αυτό είναι κάτι το οποίο καθιερώθηκε το 2003 και πραγματικά είναι πεπαλαιωμένο. Είναι στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν πια και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ε, νέα ανώτατα όρια αλληλευτικής ικανότητας ε, με βάση τα σημερινά στοιχεία και τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να εφαρμόσουν τις μεταβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις να έχουν ένα ανώτατο όριο αλληλευτικής ικανότητας ε, το οποίο να είναι χαμηλότερο από το σημερινό. Και σίγουρα να μην χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του διότι είναι πράγματι πεπαλαιωμένα. Επίση, πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κύριο Χάρτστον και άλλοι βουλευτέ, ότι μόνο οι ενεργοί αλληλεί θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να λάβουν ε, δικαιώματα αλληλεία ή παραχωρήσει, ώστε να μην έχουμε την δυνατότητα οι τράπεζε ε, ή ε, δίθεν καπετάνοι να έχουν τέτοια δικαιώματα. Ευχαριστώ. Και τελευταίος μιλητή ο κύριο Μιλάνα. Απάτε, Εισαγωγικά να πω ότι το να αντιμετωπίσει κανεί το θέμα της μεταρρύθμισης με τον τρόπο που το κάνουμε, τμηματικά δηλαδή είναι κουραστικό και θα μας αποτρέψει να δούμε συνολικά οργανικά το θέμα. Το σύνολο των αποφάσεων τις οποίες καλούμεθα να πάρουμε για κάθε κατάσταση, για κάθε θέμα αν θέλετε, μεταφερόμενα δικαιώματα, βιοπικιλότητα. Ο τρόπος που συζητάμε ε, δεν θα μας δώσει, θα έλεγα, μια συνολική ιδέα για το που θέλουμε να πάμε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε το καθήκον σαν Επιτροπή να αποδείξουμε ότι η εφαρμογή της αρχής που περιβάλλεται στην ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποτελεσματική. Δεν μπορεί να μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο είναι αυτό που θα μας υποδείξει την εναλλακτική λύση. Αυτό δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Δεν είμαι διόλου πεπισμένος ότι η εφαρμογή αυτής της νέας μεθοδολογίας, σε εισαγωγικά νέας, θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δηλαδή την μείωση της αλλιευτικής δραστηριότητας και δεν έχει αποδειχθεί αν είναι εφικτή να υπάρξει μέσω της οργάνωσης της αγοράς που προτείνει η Επιτροπή. Και στην ουσία πρόκειται και μία άρνηση της πολιτικής που ακολουθούμε μέχρι τώρα, γιατί αφήνουμε στην αγορά αποκλειστικά την ικανότητα να ορίσει τα πράγματα. Αυτό είναι παράλογο. Εγώ είμαι σε εισαγωγικά φιλελεύθερος, αν θέλετε, πολιτιστικά. Αλλά ανάμεσα στο να είναι κανείς φιλελεύθερος από τη μία και να επιτρέπει από την άλλη ότι μπορεί να εκχωριστεί μια, να εκχωρηθεί συγγνώμη, μια τέτοια ουσιαστική πηγή πλούτου και φυσική πηγή πλούτου, αυτό είναι παράλογο, είναι μια τρέλα. Γιατί στην ουσία με τις προτάσεις σας οι θεσμοί χάνουν τον έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών. Εγώ δεν είμαι ε, τόσο απεσιόδοξος και δεν θα πω ότι επέρχεται πάρα πολύ μεγάλη υπερσυγκέντρωση κτλ. Κοιτάξτε, αν δεν αλλάξουμε τα πράγματα, έτσι και αλλιώς τα δικαιώματα αυτά δεν θα κοστίζουν τίποτα, δεν θα έχουν αξία γιατί εξαρδούνται τα αλλιεύματα. Γι' αυτό είπα ότι το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι πια πρότυπο Ιζαμπέλ, γιατί το πρότυπο αυτό δεν δίνει απαντήσεις στα δικά μας προβλήματα το MSY δεν είναι επίκαιρο. Θα τα δούμε αυτά όταν τα συζητήσουμε αναλυτικά. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε οικοσυστημικά, δηλαδή αντί να παρεμβαίνουμε επί της μεθοδολογίας της αλληλείας, θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να δούμε τι δυνατότητες έχει η θάλασσα να παράγει περισσότερο. Αυτό σημαίνει άλλου είδους μεταρρύθμιση ενώ εμείς αυτό που κάνουμε είναι να φωτοτυπούμε την προηγούμενη μεταρρύθμιση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν είναι αποδεδειγμένη η μείωση της αλλιευτικής δραστηριότητας μέσω της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα συμφωνήσω, ε, κοιτάξτε αν συζητάμε επί εθελοντικής βάσεως, τι, τι συζητάμε. Στη Δανία σαν παράδειγμα τι γίνεται. Αν η επιλογή είναι επί εθελοντικής βάσεως, ας το βγάλουμε αυτό από τη μεταρρύθμιση, γιατί οι χώρες χωρίς κανόνες θα προχωρήσουν και οι χώρες οι, οποίοι θέλουν, οι οποίες θέλουν να επιβάλλουν κανόνες θα το κάνουν εις βάρος τους. Ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει, ένα τρίτο στοιχείο ο πρόεδρος μου λέει να πάω γρήγορα. Πράγματι εμείς σαν Ευρώπη λειτουργούμε με διαφορετικό τρόπο. Ξέρουμε όμως παράλληλα ότι τα μισά λιεύματα δεν ε, περιορίζονται από ποσοστώσεις. Ξέρουμε ότι στο βορρά τα πάντα είναι οι ποσοστώσεις, ενώ οι 600 ε, ποικιλίε ψαριού στην Μεσόγειο δεν υφίστανται καμία μορφή περιορισμού μέσω ποσοστώσεων. Οπότε πώς θα ρυθμίσουμε το σύστημα δηλαδή, πώς το βλέπετε αυτό. Νομίζω ότι οι συζητήσεις μας θα πρέπει να οργανηθούν πρόεδρο, ε, πρόεδρε με διαφορετικό τρόπο γιατί αυτή η αποσπασματικοποίηση της μεταρρύθμισης δεν μας οδηγεί πουθενά σαν κοινοβούλιο. Και σύν της άλλης έχω βαρεθεί γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά που δεν υπάρχει κάτι, που υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά έρχεται στο κοινοβούλιο και λέει πείτε μας ε, την εναλλακτική λύση. Κοιτάξτε το εκτελεστικό όργανο εσείς είσαστε, δεν είμαστε εμείς. Δεν έχουμε εμείς την ομοθετική πρωτοβουλία, εσείς την έχετε την νομοθετική πρωτοβουλία, εσείς πρέπει να κάνετε αποτελεσματικές προτάσεις, είναι εν πάση περιπτώσει δική σας ευθύνη και πρέπει να την αναλάβετε. Ευχαριστώ. Θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά όταν παρουσιαστεί και το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει μια σύντομη παρακαλώ παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα αρνητικά σχόλια, γιατί έγινε κάποια θετικά σχόλια για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θα απαντήσω στις επικρίσεις ή στις ε, ερωτήσεις. Ε, κύριε Καντέκ, Ήσταν πολύ επικριτικό κατά τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε το κριτήριο των 12 μέτρων ε, και το γεγονό ότι εφαρμόζεται σχεδόν σε όλου ε, οι μετεβάσιμε ε, αυτέ οι ελευτικές παρατηρήσει δεν ισχύει. Είδαμε τα στατιστικά στοιχεία και ακόμη και με το κριτήριο των 12 μέτρων, σε πολύ λίγα σκάφη του ελευτικού στόλου εφαρμόζονται αυτά τα TFC. Ακόμη και για, για την αερία ανοιχτή θάλασσα είναι πολύ μικρό το ποσοστό για το οποίο εφαρμόζονται τα TFC δεν σημαίνει κατά ανάγκη το κριτήριο των 12 μέτρων θα γενικεύσει την χρήση των TFC. Υπάρχουν κάποια θεμελιώδη ζητήματα και κάποια ε, δευτερεύοντα ζητήματα. Τώρα, για το κατά πόσο το κριτήριο των 12 μέτρων είναι το καλύτερο, αυτό είναι τεχνικό περισσότερο ζήτημα, δεν είναι ζήτημα αρχή. Θέμα αρχή για, την, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να βρούμε ένα σύστημα που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επιλύσουν με αποτελεσματικό τρόπο και ε, κατά προτίμηση με χαμηλό κόστος το πρόβλημα της, ε, του πλονάζοντος δυναμικού, της υπερπλεονάζουσας ελευτικής ικανότητας. Αυτό είναι το ζήτημα αρχής και το ζητούμενο. Για τα τεχνικά θα δούμε. Επαναλαμβάνω, η πρόταση προβλέπει ε, περιορισμούς από τα κράτη-μέλη για να αναχαιτιστεί το πρόβλημα της συγκέντρωσης, ενδεχομένως με ρήτρες διασφάλισης. Έχουμε πολλούς ελεύθερικους ε, κλάδους ε, στην Ευρώπη με υψηλό βαθμό συγκέντρωση και κανένας ε, δεν ε, διαρριγνεί τα μάτια του και δεν διαμαρτύρεται ότι είναι αρνητική αυτή η συγκέντρωση. Ακόμη και πέραν των TFC υπάρχουν ήδη συγκεντρώσεις μέσω των επενδύσεων που γίνονται από ορισμένε επιχειρήσει άλλε και από ορισμένε χώρε άλλε και κανένα διαμαρτύρεται για τη συγκέντρωση αυτή. Επαναλαμβάνω, το θέμα τη συγκέντρωση είναι θέμα επενδύσεων. Και δύο επιχειρήματα μου έρχονται εδώ. Αυτό ήδη ισχύει. Για να υπάρχουν επενδύσεις και να υπάρχει συγκέντρωση επιχειρηματική δεν χρειαζόμαστε καν τι μεταβιβάσιμε αλληλευτικέ παραχωρήσεις. Τώρα, αν θεωρείτε ότι είναι κίνδυνο να γίνονται επενδύσεις από τη μια χώρα στην άλλη, τότε καλώ ήρθατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο να σα πω. Ο κύριος Φεραίρα έδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πού υπάρχει το πλεονάζον δυναμικό, υπερβάλλουσα αλληλευτική ικανότητα. Αυτό προσπαθούμε να ε, ελέγξουμε από το 2003. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπονεί ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του άρθρου 11 του βασικού κανονισμού, δηλαδή για την εφαρμογή τη πολιτική μα στον αλληλευτικό στόλο. Αυτή η έκθεση γίνεται ετησίω με βάση τι εθνικέ εκθέσει. Και η προσωπική μου απογοήτευση και ο εκνευρισμό για την ειδική μου ευθύνη είναι ότι όταν τα κράτη-μέλη μα στέλνουν τι εθνικέ του εκθέσει, Σχεδόν σε καμία έκθεση δεν υπάρχει αποτίμηση του πλεονάζοντος δυναμικού και το πού υπάρχει αυτή η πλεονάζουσα ικανότητα. Είναι κάτι που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κάνουν. Δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κράτη-μέλη δεν καταφέρουν να αποτιμήσουν αυτό το πλεονάζον δυναμικό. Τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν ε, τα στοιχεία αυτά, δεν μπορούν να αναλύσουν με λογικό τρόπο το ζήτημα του υπερβάλλοντος ελευτικού δυναμικού. Κανένα κράτος δεν μας έχει δώσει ξεκάθαρη απάντηση για αυτό το ερώτημα που έχουμε δώσει και εδώ ε, και νέα χρόνια αυτό το ζητούμε. Τώρα, αν ε, θα εξοβελιστούν ε, από το παιχνίδι τα ελευθερικά σκάφη που έχουν περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα και θα παραμείνουν αυτοί που έχουν πιο οικονομικά αλλά λιγότερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Τι να σας πω, ε, θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία κυρίως στους αλληλείς που ε, πραγματοποιούν βιώσιμη αλία και με σωστά δίχτυα. για να αποφύγουμε τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Αυτό όμως θα το θα το φροντίσουμε μέσω του συστήματος Τίποτα βέβαια δεν εξασφαλίζει τη μείωση του πλεονάζοντος δυναμικού. Ο κύριος Μιλάνε είπε ότι δεν έχουμε αποδείξει ότι θα λειτουργήσει το σύστημα. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ένα σύστημα που δεν έχει ουδέποτε εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει. Αυτό που μπορούμε να αποδείξουμε είναι ότι στι χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και στι χώρε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει εφαρμοστεί το σύστημα υπήρχαν αποτελέσματα. Το σύστημα λειτουργήσε. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε. Και ταυτόχρονα αυτό που μπορούμε να αποδείξουμε ακόμη καλύτερα είναι ότι το ισχύον σύστημα είναι τελείω αναποτελεσματικό. Μπορεί κανεί να επικρίνει τις ε, μεταβάσιμες ελευτικές παραχωρήσεις. Σίγουρα δεν είναι πανάκια, είμαστε οι πρώτοι που το δηλώνουμε. Αλλά όπως είπε και η Επίτροπος Ελίας, αν έχετε άλλη εναλλακτική λύση, πείτε το μας. Εγώ δεν έχω ακούσει όμως καμία άλλη εναλλακτική πρόταση. Οπότε η συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι η συζήτηση μεταξύ τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι μεταβάσιμε ελευλευτικέ παραχωρήσει αλληλευτικές μέχρι τώρα κατάσταση. Γιατί ή του Στάτου Κβό, μέχρι τώρα κατασταση Γιατί εναλλακτική πρόταση δεν έχει υποβληθεί από κανέναν. Αυτό που είναι πασιφανές πια είναι ότι το ισχύο σύστημα δεν λειτουργεί. Η κυρία Μπιλμπά μας ζήτησε ένα, μια πλήρη απεικόνηση της κατάστασης. Όπως είπα, τα κράτη αδυνατούν να κάνουν κάτι τέτοιο από μόνα τους. Τώρα, ένας από τους λόγους για τους οποίους προτείνουμε το νέο σύστημα είναι ότι για τους λόγους που σας εξηγήσαμε και αν θέλετε μπορούμε να σας τους ξαναεξηγήσουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι και οι επιδοτήσει για τον παραπλησμό δεν λειτουργήσαν. Γιατί ε, ήταν πολύ μεγάλα κονδύλια, πολύ ψηλά κονδύλια των Ευρωπαίων φορολογούμενων και τελικά το πρόβλημα παρέμεινε ανεπίλητο. Η κυρία Λόβιν μας, μας ρώτησε γιατί θα πρέπει η κατανομή να γίνει με βάση τα ιστορικά ελιεύματα. Καμία υποχρέωση. Όπως είπα και εγώ, το σύστημα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν με κυρίαρχο τρόπο τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν για να κατανείμουν τα ελευτικά δικαιώματα μεταξύ των αλλιέων τους. Αν λοιπόν μια χώρα θέλει στην κατανομή να ευνοήσει συγκεκριμένες δραστηριότητε, μπορεί κάλλιστα να το κάνει. Εμείς δεν εμποδίζουμε κανέναν το κράτος μέρος. Και για το ότι είναι υπερβολική η διάρκεια των 15 ετών. Αυτά είναι τεχνικά θέματα, επαναλαμβάνω. Και για αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να μαλώσουμε αν κάποιο ε, πιστεύει και αποδείξει ότι μια άλλη διάρκεια είναι πιο πρόσφορη, πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα όρια του δυναμικού, φαίνεται ότι είναι παροχημένα. Για μας το θέμα είναι αν τα συστήματα αυτά εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και αν γίνει ε, η αναθεώρηση υπάρχει κάποια χρησιμότητα. Αυτά τα όρια ε, της γίνονται σεβαστά από όλα τα κράτη-μέλη, οπότε πρόβλημα δεν υπάρχει. Ακόμη ε, και τα κράτη-μέλη είναι κατά μέσο 10% κάτω από τα όρια, οπότε τα όρια αυτά δεν περιορίζουν κανέναν. <clears throat> τα όρια αυτά είναι, προϋποθέτουν έναν διοικητικό φόρτο χωρίς αποτέλεσμα. Έχει νόημα μια τέτοια πολιτική. Όχι, γι' αυτό και αν ε, εφαρμόσουμε το σύστημα των μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων, δεν θα συνεχιστεί το προηγούμενο σύστημα. Ο κύριος Μιλάνα ρώτησε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το, θέμα, αυτό το σύστημα των TFC στη Μεσόγειο. Το σύστημα δεν θα ισχύσει μόνο με βάση τις ποσοστώσεις αλλά και με βάση την αλληλευτική προσπάθεια. Και στον κανονισμό για τη Μεσόγειο προβλέπεται τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν σχέδια διαχείρισης με βάση την παράμετρο αλληλευτική προσπάθεια και τη στιγμή που θα εφαρμοστούν τα σχέδια διαχείρισης στη Μεσόγειο και όταν θα προσδιοριστούν αυτές οι προσπάθειες, οι ποσοστός αλληλευτικής προσπάθειας, τότε μπορεί να ε, περιληφθούν στο σύστημα των ε, μεταβιβάσιμων αλληλευτικών παραχωρήσεων. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Η κυρία Ρόντουστ για να δευτερολογήσει θέλει κάποια διευκρίνηση. Äh, ήθελα να αναφερθώ στις ε, διάφορες παρεμβάσεις, αλλά εντάξει δεν χρειάζεται να το κάνω. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι ένα πράγμα ε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Να πούμε ότι δεν ε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει γρήγορα να βρούμε μία λύση. Άκουσα πολλά, δεν άκουσα καμία πρόταση λύσης. Σας παρακαλώ λοιπόν να καθίσετε, να, γράψετε, να καταγράψετε ιδέες. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μέσο στα χέρια μας. Νωρίτερα η Κομισιόν τα έκανε όλα μόνη της. Ε, τώρα έχουμε την συναπόφαση. Τώρα καθόμαστε και εμεί στο τραπέζι με ίσα δικαιώματα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο να δημιουργηθούν κίνητρα Ήδη έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές. Ε, χρήσιμο θα είναι λοιπόν να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση. Το να πούμε ότι δεν υπάρχει λύση δεν είναι λύση. Ε, χρειαζόμαστε μια τέτοια λύση, χρειάζομαι τις προτάσεις σας ε, και ε, το να ε, φοβούμαστε να κάνουμε κάτι δεν ε, είναι σωστό τα, μπορούν κάλλιστα να ε, δημιουργηθούν τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης, ε, η επίκριση ότι εδώ πέρα ασχολούμαστε μόνο με κάποιες λεπτομέρειες του θέματος ε, δεν ισχύει. Ή να σας το πω αλλιώς, εγώ χρειάζομαι να το κάνω, να εξετάσω το θέμα σε φέτες. Ε, δεν έχω ξεχάσει το σύνολο, αλλά ε, θέλω να συζητήσουμε ενδελεχώς κάθε κομμάτι του βασικού κανονισμού και στο τέλος ε, θα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε μια αποτελεσματική δέσμη προς όφελος των αλλιέων, των ανθρώπων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Pasamos Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το 25 αντί για το 24, γιατί αλλάξαμε τη σειρά των σημείων και θα περάσουμε στο σημείο 25. Μας έμειναν τρία τέταρτα για τρία ζητήματα. Γι' αυτό και θέρμο παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας παρουσιάσει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Thank you, Chair. Uh, Johan uh, representing the... Ευχαριστώ. Ε, Προσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Θα σας παρουσιάσω συνοπτικά τις βασικές γραμμές των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πλαίσιο 14 με 20 εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, τι είναι αυτό το πολιετές πλαίσιο. Και δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στο νέο νομικό πλαίσιο με το οποίο εργαζόμεθα σίγουρα σήμερα. Το MFF είναι ένας πίνακας ουσιαστικά που περιλαμβάνει τα ανώτατα όρια δαπάνης, τα, τα επιτρεπόμενα όρια δαπάνης, κατέτος και τομέα δαπάνης. Πρόκειται για ένα πίνακα σύμφωνα με τον οποίο θα κινηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός. Ο πίνακα συνοδεύεται από ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναθεωρείται ο πίνακας, κάτω από ποιες συνθήκες και πώς τα όρια που περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτά μπορεί να ξεπεραστούν κάτω από πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Γιατί είναι αυτό το MFF τόσο σημαντικό είναι αν θέλετε το θεμέλιο που επιτρέπει το, ε, <clears throat> την πολυετή οικονομική μορφή προγραμματισμού. Θέτει το πλαίσιο έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν αρκετά χρόνια πριν πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα, πόσα είναι τα ανώτατα όρια και τι μπορεί να περιμένουν. Δεύτερον, το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει τη λεγόμενη δημοσιονομική ειρήνη από την αρχή της ισχύω των πλαισίων αυτών από το 1998 και μετά, ποτέ δεν υπήρξε μια άκερη υιοθέτηση του προϋπολογισμού ή με μεγάλη καθυστέρηση. Το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τη συνδύσικη της Λισαβόνας λέει το εξής. Μέχρι τώρα το πολιετές αυτό πλαίσιο ήταν τμήμα μιας διοργανικής συμφωνίας ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αυτό έχει αλλάξει πλέον. Το άρθρο 312 ε, της Συνθήκης της Λισαβόνας εισάγει έναν κανονισμό, έναν κανονισμό του Συμβουλίου, ο οποίος θα υιοθετείται ομόφωνα μεν, αλλά, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερη καινοτομία, σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφορά τη χρηματοδοτική πλευρά του προϋπολογισμού. Το Σημείο 4 εισάγει τη δυνατότητα των λεγόμενων εφαρμοστικών κανονισμών. Μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε απλά να γνωμοδοτήσει επί, του, επί της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού, ενώ αυτός ο κανονισμός του Συμβουλίου θα υποβάλλεται προς έγκριση και στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της στις 29 Ιουνίου, ο πρόεδρος Μπαρόσο τις χαρακτήρισε τις προτάσει αυτές φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τα δύο αυτά στοιχεία της πρότασης. Πρώτον, γιατί η πρότασή μας είναι ρεαλιστική. Η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε είναι η εξής. Να αναφέρω τρία στοιχεία. Το υπάρχον πλαίσιο συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο 2007-2013. Ένα του γενικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του συνόλου της οικονομίας μας. Λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε, έχει αυξηθεί στο 1,12%. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ένα μεγαλύτερο κομμάτι των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας από ό,τι προβλέπαμε στο παρελθόν. Δεύτερο στοιχείο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα συμπεράσματα της Επιτροπής της Αρμόδιας του Κοινοβουλίου που υιοθέτησε την έκθεση της πέρυσι λέγοντας ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα πρέπει να είναι κάτω από το 1,11% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Τρίτο θεμέλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παρουσιάζει την πρότασή της είναι το ότι γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σκληρά σε επίπεδο δημοσιονομικής πειθαρχία και έχουν διευκρινίσει ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση ένα ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ανώτερο του 1%. Πώς θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τετραγωνίσουμε τον κύκλο αυτών των διαφορετικών απόψεων. Το κάναμε αυτό αντιστρέφοντας, επιστρέφοντας στη συμφωνία του 2005 Συμβουλίου Κοινοβουλίου και θέτοντας αν θέλετε την πρότασή μας στο 1,05%. Ταυτόσιμο δηλαδή με τη συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου το 2005. Αλλά παρόλα αυτά ρίξαμε γέφυρες και προς το Κοινοβούλιο και προς το Συμβούλιο. Προς το Κοινοβούλιο ρίξαμε γέφυρες διευκρινίζοντας ότι εκτός του 1,05 έχουμε ένα επιπλέον δυνατόν ποσό 0,06% πιθανής δαπάνης που συνολικά μας φτάνει στο 1,11%. Τον αριθμό δηλαδή στον οποίο αναφέρθηκε η Επιτροπή Σούρε. Αυτό το 1,05% είναι για τις πιστώσεις υποχρεώσεων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάσαμε ένα όριο για τις πιστώσεις πληρωμών, αντίστοιχο με 1,00. Και αυτή είναι η γέφυρα την οποία, αν θέλετε, στέλνουμε, ρίχνουμε προς τους πιο αυστηρούς δημοσιονομικά η πρότασή μας είναι αρκετά φιλόδοξη, όχι μόνο ρεαλιστική όμως, γιατί ακριβώς μέσα σε αυτό το 1,05% έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε τις δύο πιο μεγάλες δαπάνες, την ΚΑΠ από τη μία και την συνοχή από την άλλη. Μέσω της σταθεροποίησης αυτών των δύο πυλώνων μέχρι το 2000, από το 2013, ε, θα έλεγα ανοίξαμε ένα περιθώριο έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες στοχευμένες αυξήσεις σε ορισμένες πολιτικές μετά το 2013. Δεύτερον, και σχετικά με τα στοιχεία εκτός του 0,06%, ε, προτείνουμε ακόμα περισσότερη ευελιξία, σημαντική για το Κοινοβούλιο, προτείνουμε κάποια επιπλέον ποσά, προτείνουμε ένα νέο μέσο ευελιξίας για τις αγροτικές τιμές, και προτείνουμε επίσης να μετακινήσουμε εκτός του πλαισίου τα δύο βασικά προγράμματα, τα οποία είναι το GMES και το ITER. E Αυτά είναι λοιπόν τα θεμέλια πάνω στα οποία βασίζεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κλείνοντας, Πρόεδρε, θα σας περιγράψω το τι πρέπει να πετύχουμε. Κοιτάξτε, κλείστε παρακαλώ γιατί υπάρχει και ένα συνάδελφό σα που θέλει το λόγο, δεν έχουμε πολλή ώρα. Θα είμαι πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει αυτός ο κανονισμός MFF να υιοθετηθεί με ομοφωνία στο Συμβούλιο και επίσης στο Κοινοβούλιο, διότι αυτό θα επιτρέψει το 2013 στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ξεκινήσουν τις διάφορες τομεακές δράσεις, ώστε όλα να τεθούν σε σχητη 1 1η Ιανουαρίου του 2014. Κύριε Τζόνσον, παρακαλώ, χρόνο φίδου. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρει την Επιτροπή μας οι δαπάνες ε, στον ε, τομέα της αλίας, ε, το πολιετές πλαίσιο περιέχει πέντε τίτλους, αυτό λέει η πρόταση και οι δαπάνες βρίσκονται στον τίτλο 2. Ο τίτλος 2 λέγεται «Βιώσιμη ανάπτυξη φυσική πόρη». Η Άλλη δαπάνη που αναφέρεται εδώ πέρα είναι της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής, καθώς και η ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και περιβαλλοντικές δαπάνες ε, και δαπάνες για τη βελτίωση του κλίματος. Η συμπερίληψή μας στον τίτλο 2 είναι παρόμοια με την παρούσα κατάσταση και εκεί βλέπουμε τις δαπάνες για τις παρούσες για το παρόν ε, πολιετές πλαίσιο που θα λήξει το 2013. Οι στο στόχο έχουν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τη Ευρώπη 2020. Όσον αφορά λοιπόν τα θαλάσσιε υποθέσεις και την αλληλεία, ε, θα συμβάλλουμε ε, έτσι στην ανάπτυξη και καλύτερη απόδοση, όπως επίσης στη δημιουργία θέσεων εργασίας να αναφερθώ στα ποσά για τα οποία μιλάμε, διότι αυτό μας ενδιαφέρει. Το συνολικό ποσό για ε, θαλάσσιες υποθέσεις και αλληλεία, το ποσό είναι 7 δισεκατομμύρια, 536 εκατομμύρια. Ε, αυτό αποτελεί το 0,65% των συνολικών δαπανών. Τι σημαίνει αυτό, ότι ουσιαστικά ξεκινάμε με ένα ε, δισεκατομμύριο ε, δισεκατομμύριο το πρώτο έτος και το 2020 καταλήγουμε με ένα δισεκατομμύριο 550.000. Ε, ο φάκελος αυτός ε, καλύπτει όλους τους τομείς με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον έλεγχο της αλίας που καλύπτεται από διαφορετικό φάκελο για τις υπηρεσίες. Να μην μακρηγορήσω, να κλείσω λέγοντας ότι προτείνουμε ένα όργανο ε, για την πιστοποίηση. Έχουμε ενοποιήσει λοιπόν πέντε νομικές βάσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Θαλάσσης και Αλληλείας ε, το οποίο θα είναι ο απόγονος του EFF, του IFP, του μέσου για τις δαπάνες για την αγορά, καθώς και για το μέσο για τις πιο απόμακρες περιοχές. Όσον αφορά την απλοποίηση, το άλλο που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να απλοποιήσουμε το σύστημα παράδοσης, ώστε η ζωή να γίνει πιο εύκολη για τα κράτη-μέλη και για τους δικαιούχους όμως. Και τέλος, για να έχουμε πλήρη εικόνα για τις δαπάνες ε, για τη θάλασσα και την αλληλεία, είναι απαραίτητο να, πάρουμε, να λάβουμε υπόψη και ε, αυτά που έχουμε ε, βάλει κατά μέρο για τις περιφερειακές, ε, περιφερειακές οργανώσεις καθώ καθώς και για τις ε, συμφωνίες βιώσιμη ε, που είναι όπως οι αλληλευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και μιλάμε για 968, εκατομμύρια. Ο κύριος Φερέρα, παρακαλώ να τηρήσετε τις υποσχέσεις σα. Υποσχέθηκα στον κύριο Κάλεχερ ότι δεν θα πω τίποτα για το σημείο αυτό θα έχουμε ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε σε άλλη συνεδρίες. Ευχαριστούμε κύριε Φερέιρα. Άλλε παρεμβάσει δεν έχουμε. Περάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη και πάλι είμαστε υπατμών. Το σημείο 24. Ορισμένα μέτρα κατά το χωρών οι οποίε επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμη αλία με στόχο τη διατήρηση των ηχθείων αποθεμάτων. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σύντομη παρουσίαση θα έχουμε και ανταλλαγή απόψεων. Ο, παρακαλώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Εν συντομία θα σας παρουσιάσω την πρόταση. Ο λόγος της υποβολής πρότασης ε, ήταν ε, η κατάσταση αποθεμάτων ε, σκουμπριού στο Βόρειο Ατλαντικό. Γι' αυτό και θεσπίστηκαν τα σχετικά μέτρα. Είναι πιο σημαντικό ε, αλληλευτικό απόθεμα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχή Νορβηγίας, Φερών και Ισλανδίας. Εδώ και δύο χρόνια δεν καταφέραμε να καταλήξουμε συμφωνία για κοινή διαχείριση του ελευτικού υποθέματος σκουμπριού, κάτι που δημιουργεί σοβαρές ε, ανησυχίες για την βιωσιμότητα. Από μόνη της Ισλανδία, για παράδειγμα, έχει αλλιεύσει το ένα περίπου τέταρτο των αλλιευμάτων ε, με βάση το λογικό κατά τη γνώμη των επιστημόνων πέρυσι, το λογικό αλλιεύμα. Αυτά τα ελληνικά αποθέματα θα πρέπει να τύχουν κοινή διαχείριση, καλόπιστη κοινή διαχείριση μεταξύ των ε, παράκτιων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, τη Ισλανδία και άλλων. Στόχο τη πρότασή μα λοιπόν ε, είναι να εξασφαλίσουμε την αηφορία, την βιωσιμότητα, τη βιώσιμη εκμετάλλευση αυτών των αλληλευτικών πόρων, αυτών των ηχθιαποθεμάτων. Και επίσης ε, ε, να αποφύγουμε την τη μονόπλευρη δράση, να δημιουργήσουμε κίνητρα για κοινή διαχείριση και συνεργασία μεταξύ των παράκτων χωρών. Αυτό είναι ο στόχος της πρότασης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 και αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τέτοιας έλλειψης συνεργασίας. Η πρόταση κανονισμού στη συνέχεια προσδιορίζει τις χώρες κατά, τις οποίες, ε, κατά των οποίων μπορούν να ληφθούν τέτοια μέτρα Πρόκειται για χώρε που επιτρέπουν τη διεξαγωγή μη βιώσιμη αλίας. Υπό δύο όρου γίνεται η λήψη των μέτρων. Καταρχήν ε, ε, έλλειψη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον κίνδυνος αυτά τα μέτρα διαχείρισης που λαμβάνει η μονόπλευρα η χώρα αυτή να διακυβεύουν τη βιωσιμότητα των ηχθειαποθεμάτων. Ο υπόλοιπο κανονισμό προβλέπει μία σειρά μέτρων ε, που μπορεί να ε, ληφθούν με βάση τον κανονισμό για την άναρχη παράνομη και αδήλωτη αλία. Υπάρχει δηλαδή σχετική νομοθεσία αφορά τον προσδιορισμό των χωρών που επιτρέπουν μη βιώσιμη αλία και ε, ως μέτρα προβλέπει την ε, μείωση των εισαγωγών, κάποια μέτρα εμπορικά και περιορισμό παροχής υπηρεσιών όπως είναι η πρόσβαση στα λιμάνια. Φυσικά αυτά τα μέτρα όπως αναφέρεται στον κανονισμό ρητά θα πρέπει να είναι συμβατά με τις διεθνείς συμφωνίες, ιδιαίτερα με την ΚΑΤ. Θα πρέπει να, να μην ε, είναι διακριτικά δηλαδή να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ κοινοτικών και εξωκοινοτικών χωρών ε, και θα πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχε προδιαγραφές ε, και στους κοινοτικού και στους εξοκοινοτικού αλληλείς. Και σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε για την ε, λήψη αυτών των μέτρων, οι διαδικασίε αυτέ μιλάνονται από την ανάγκη δίκη αυτές εμπνέονται από την ανάγκη δικη και άμεσης δράσης. Και εδώ η ταχύτητα είναι ζωτική σημασία, γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε από θέματα που κινδυνεύουν. Υπάρχει υποχρέωση κοινοποίηση της χώρας και προβλέπεται διαδικασία που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει εφαρμοστικά μέτρα, εφαρμοστικές πράξεις, συγγνώμη, προκειμένου να εφαρμόσει τα μέτρα που προσδιορίζονται ρητά στον κανονισμό. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο προσδιορίζει τα κριτήρια, τον τρόπο εφαρμογής σε μεμονωμένες καταστάσεις και θα πρέπει αυτό να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται με συνοπτικό και ταχύ τρόπο και πιστεύουμε ότι η πρόταση το επιτρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω γιατί είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή της πρότασης. Ε, ήταν άλλωστε πρωτοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διέβλεψε τον κίνδυνο μιας τέτοιας πρακτικής για τη διατήρηση των ηχθείων αποθεμάτων και επισήμανε την ανάγκη λήψη κάποιων μέτρων. Φυσικά είπαμε θα πρέπει να τηρήσουμε το, τις διεθνείς νομοθεσίες και φυσικά εδώ η λέξη κλειδί είναι βιωσιμότητα, βιώσιμη αλεία, αηφορία της αλείας. Είχαμε την εμπειρία και από τον αποδεκατισμό των ηχθιαποθεμάτων προσφυγακίου εξαιτία έλλειψη συμφωνία μεταξύ των παράκτιων χωρών. Πραγματικά θα πρέπει να αποφύγουμε αντίστοιχη κατάσταση και σε άλλα ηχθιαποθέματα. Τώρα για τον κανονισμό. Αν ε, εφαρμοστεί αυτή η ανακοίνωση, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα αν δεν ε, έχουμε σοβαρές εξηγήσεις ή ε, ριζική μεταρρύθμιση του άρθρου 4. Το άρθρο 4 επιβάλλει ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ε, σε προϊόντα ή σε ε, ψάρια που προέρχονται από το συγκεκριμένο ηχθιαπόθεμα. Αυτό να το τονίσουμε, γιατί στο παρελθόν είχαμε το προσφυγά και τώρα έχουμε το σκουμπρί. Αλλά νομίζω ότι μια, ένας τέτοιος περιορισμός δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Επίσης προβλέπει ποσοτικούς περιορισμούς ε, εισαγωγής ε, ε, όχι, των ε, συγκεκριμένων ψαριών και των συναφών ειδών. Τι θα πει συναφών ειδών, θα πρέπει να το προσδιορίσουμε και αυτό. Στην επόμενη συνεδρίαση λοιπόν θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτά τα σημεία και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να πούμε ότι η παράγραφος Γ διαγράφεται και αναδιατυπώνεται η παράγραφος Δέλτα. Αυτά προς το παρόν γενικά. Τώρα, ως προς την επιβολή ε, ποσοτικών περιορισμών για την εισαγωγή στην Ένωση ε, ψαριών και Λιευτικών προϊόντων, οποιοδήποτε είδος που προέρχεται από τη χώρα αυτή που επιτρέπει μη βιώσιμη αλληλεία και όχι μόνο συγκεκριμένων αλληλευτικών ειδών. Και γιατί το λέω, γιατί αν περιοριστούμε σε συγκεκριμένα αλληλευτικά είδη που υπεραλλιεύονται, δεν θα πάμε πουθενά, γιατί το 95-98% των προστατευμένων ειδών που μιλάμε δεν έρχονται καν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1% ποια διαφορά. 1-2%. Ίσως αυτή είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ίσως προτρέχω εδώ και προεξοφλώ την οριστική μορφή της πρότασης. Περιμένουμε ε, νέα συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, ε, το γεγονός ότι έχουμε διαπραγματεύσει για το θέμα αυτό με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευελπισώντα ότι θα το διεκπαιρεώσουμε τον Ιούνιο-Ιούλιο, πιστεύω ότι και μόνο, από αυτό, και μόνο το αυτό το γεγονός θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, να μην κατανομάσουμε συγκεκριμένε χώρε. Σε ό,τι αφορά τι τελευταίε πληροφορίε που είχα το πρωί, φαίνεται ότι η Ισλανδία το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα και φαίνεται ότι ήδη διαφαίνεται κάποια πρόοδο. Ό,τι αφορά τι Φερόε όμω, εκεί υπάρχει μια διαλαξία Και μάλιστα προβλέπουν ποσοστώσεις που είναι πολύ ψηλότερες από τις δικές μας. Και χρησιμοποιούν ολόκληρα πλοία εργοστάσια, μεταποιώντας το προϊόν επιτόπου. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε ούτε δείγμα ψαριού για τα παράκτια κράτη. Και η Νορβηγία βέβαια ήταν συνυπεύθυνη για το θέμα αυτό και η Φερόες και η Ισλανδία, αλλά τουλάχιστον η Ισλανδία δείχνει μια επιθυμία πρόοδου. Εν ολίγης, ε, οι επιστήμονες μας είπαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, λέει ότι οι εμπειρογνώμονες ε, το τόνισαν. Πέρυσι αλλιεύθηκε ένα εκατομμύριο τόνι, ενώ για το, το βιώσιμο ποσοστό είναι 650.000 τόνι. Τι σημαίνει, αποδεκατίζονται τα ήχθη αποθέματα. Βέβαια τα ψάρια δεν γνωρίζουν γεωγραφικά σύνορα. Σε λίγα χρόνια θα μεταφερθούν προς άλλα χωρικά είδωτα. Εδώ είναι πραγματικά ένας τομέας που χωρίς συνεργασία. Θέλουμε ορθολογική, ε, βιώσιμη αλία και λαμβάνοντας υπόψη και τις επερχόμενες γενιές γιατί γίνονται τεράστιες επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ιδιωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Επιτροπή, η Ένωση, το Κοινοβούλιο θέλουν να φροντίσουν τα ηχθιαποθέματα. Χρειαζόμαστε συνεργασία γι' αυτό. Διευκρίνηση όμως, η σήμερα ή αργότερα, τι ακριβώς εννοείται με το associated species, τα συναφή είδη, τα συναφή αλληλευτικά είδη. Εγώ θεωρώ ότι μιλάμε για ε, αλίευμα και αλευτικά προϊόντα οποιοδήποτε αλληλευτικού είδου που προέρχονται από τη χώρα αυτή που επιτρέπει μη βιώσιμη αλία, όχι μόνο περιορισμό σε συγκεκριμένα ελευτικά είδη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ανα πάσα στιγμή να υποβάλει νομοθετικέ προτάσει και την ευχαριστώ θερμά γιατί μερικέ φορέ ε, είμαστε αυστηροί απέναντι στην Επίτροπο και επικριτικοί απέναντι στην Επιτροπή. Στη συγκεκριμένη όμω περίπτωση έδρασε άμεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την υποστήριξη του κλάδου και την υποστήριξη της δικής μας Επιτροπής. Η κυρία Λέβεν και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, σαν σκιώδης. Δεν μπόρεσα να δω όλες τις λεπτομέρειες της πρότασης, αλλά υποστηρίζουμε γενικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε όμως να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εμβάθυνση. Κυρία Φρέκυρε, ε, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας. Ε, νομίζω ότι ο εισηγητής ε, περιέγραψε τα, τις πολιτικές δυνάμεις πίσω από αυτό. Θα ήθελα να αναγνωρίσω την ανάγκη ότι το μέτρο αυτό θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και γι' αυτό δεν μπορεί να περιορίζεται σε κάποια είδη μόνο. Ε, πολύ ευχαρίστω ε, θα συζητήσουμε μαζί σα πώ μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό το μέτρο αυτό. Προβλέπουμε επίση μέτρα τα οποία ξεπερνάνε τι εισαγωγέ, όπω είναι η χρήση ε, λιμενικών υπηρεσιών που αποτελούν επιπλέον κίνητρο για τι χώρε αυτέ. Και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ε, ε, ένα πολύ ιδιαίτερο μέτρο, αλλά σίγουρα ε, θεωρούμε και εμείς σημαντικό το θέμα αυτό και πολύ ευχαριστώ σας συμμετάσχουμε στην επίλυσή του. Καλώς περνάμε στο επόμενο σημείο, το υπαριθμό 20. Τροποποίηση του κανονισμού 1185 του 2003 σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφου. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ πρώτα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Θεοφύλλων, δεν κάνω λάθος. Thank you, Chairman. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, δίνοντάς σας κάποιες γενικές πληροφορίες ε, για την πρόταση αυτή, την οποία υιοθετήσαμε στις 21 Νοεμβρίου 2011. Η πρόταση αυτή βασίστηκε μεταξύ άλλων ε, στον ε, μεγάλο ε, αριθμό απαντήσεων που λάβαμε σε δημόσια διαβούλευση. Λάβαμε 5.500 απαντήσεις πρόταση αυτή λοιπόν στόχο έχει να τροποποιήσει την ε, παρούσα απαγόρευση για ε, την αφαίρεση πτεριγίων καρχαρία. Ε, για να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγχυση, thinning είναι η αφαίρεση πτερυγίων του καρχαρία και κατόπιν η απόρριψη του καρχαρία στη θάλασσα. Υπάρχουν κατ' εξαίρεση οι οποίες μπορούν να εκδοθούν από ε, χώρες σημαία που επιτρέπουν μεταποίηση ε, στο σκάφος. Ε, επιτρέπουν δηλαδή την αφαίρεση του πτεριγίου εφόσον μείνει ο υπόλοιπο καρχαρίας και τον μεταποιήσουν στο πλοίο. Στην περίπτωση που επιτρέπεται τέτοια μεταποίηση υπάρχει αναλογία βάρους 5% δεν επιτρέπεται δηλαδή τα πτερίγια στο σκάφος να ξεπερνούν το 5% του βάρους ε, των ε, καρχαριών ε, που έχουν αλλιευτεί και βρίσκονται στο πλοίο. Δεν υπάρχει ενιαίο ποσοστό που να μπορεί να εφαρμοστεί για όλα τα είδη καρχαριών και τις διάφορες τεχνικές κοπής. Χρησιμοποιούνται δηλαδή διάφορες τεχνικές κατά την αποκοπή των πτερυγίων. Ε, άλλο πρόβλημα με το παρόν σύστημα που δυσκολεύει τον έλεγχο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εκφορτώσεις επιτρέπονται, ξεχωριστές εκφορτώσεις επιτρέπονται, ώστε επιτρέπεται να γίνει εκφόρτωση πτεργίων και καρχαριών σε διαφορετικά λιμάνια και ε, γι' αυτό οι επιθεωρητές θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στα ημερολόγια των πλοίων και να ε, συγκρίνουν τα στοιχεία αυτά με το θεωρητικό ε, βάρος των ζωντανών καρχαριών για να διαπιστώσουν ότι δεν έχει ξεπεραστεί το ποσοστό του 5%. Η νέα πρόταση θα εξαλείψει το πρόβλημα των ειδικών αυτών αδειών αλληλείας. Δεν θα επιτρέπεται πια επεξεργασία στο πλοίο θα πρέπει ε, οι καρχαρίες να εκφορτώνονται ε, προτού κοπούν τα πτερίγια ε, στα λιμάνια και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που μπορούν έτσι να δημιουργηθούν για τους ε, αλληλείς, για τους οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι θέματα αποθήκευσης και ασφάλειας στο πλοίο. Υπάρχει λοιπόν μια ρήτρα στη νέα πρόταση, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στο προσωπικό εν μέρη να κοπούν ε, τα, ε, πτερίγια και να διπλωθούν πάνω στο, στο ψάρι, ε, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος από ε, τα παγωμένα πτερίγια όταν ξέχουν, να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Και επίση για να λυθεί το πρόβλημα του περιορισμένου χώρου ε, πάνω στα πλοία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η συγκεκριά μα, η κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω, η απαγόρευση του φίνινγκ αυτή τη πρακτική αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφου στα χωρικά είδατα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίστηκε ελήφθη ήδη από το 2003 από το 2003 και μετά είχαμε πολλές εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο το 2006 συγκεκριμένα, που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν λαμβάνει χώρα αυτή η πρακτική της αφαίρεσης πτερυγίων καρχαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε φαίνεται ότι διαπράττουμε ένα σφάλμα. Γιατί προσπαθούμε να ρυθμίσουμε κάτι μια πρακτική που είναι ανύπαρκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, τα ίδια τα κοινωτικά θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ε, έλλειψη αυτής της πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ε, η πρακτική της αφαίρεσης ε, πτεριγιών καρχαρία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι στις ασιατικές αγορές, για παράδειγμα, για να δώσω ένα παράδειγμα, το 90% στο Χονγκ Κόνγκ των, των από των αποφορτώσεων, ε, των εκφορτώσεων γίνονται πτερυγίων καρχαρία γίνονται στο Χονγκ Κόνγκ. Και ξέρουμε ότι η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία είναι συνήθις πρακτική. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Ελευτικός ε, Στόλος δεν εφαρμόζει αυτό το φίνινγκ. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε καταδικάσει συλλήδιν το φίνινγκ. Σε πολλά επίπεδα όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, γιατί και από αυτή την άποψη ε, είναι υπερβολική, αλλά και από διοντολογικούς λόγους. Το φίνινγκ θα πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα από όλου. Αλλά επαναλαμβάνω, ο ελληνικό στόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζει πρακτική φίνινγκ. Οπότε, περί τίνο πρόκειται. Με το άρθρο 4 προβλέπεται μία εξαίρεση που επιτρέπει σε ορισμένα αλληλευτικά σκάφη με συγκεκριμένους όρους όμως που είναι πολύ αυστηροί πολύ περιορισμένα λοιπόν επιτρέπει σε ορισμένα σκάφη του Ευρωπαϊκού Ελευτικού Στόλου να κάνουν τη μεταποίηση εντός του σκάφους. Γι' αυτό ε, αφαιρούνται τα πτερίγια, ε, διαχωρίζονται από το σώμα, από τον κορμό του Καρχαρία εντός του σκάφους. Περί αυτού πρόκειται. Υπό ορου όμως πολύ λέει Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι η πρόταση ε, ανέκυψε μετά από μια διαβούλευση. Αυτή είναι η βάση για την ε, πρόταση της κατάργησης της εξαίρεσης. Τι διαβούλευση είναι αυτή όμως. Με ποιον έγινε η διαβούλευση ξέρουν οι συμμετέχοντες της διαβούλευσης περί τίνος πρόκειται είναι σαν και εμάς και είναι κατά του φίνινγκ. Γιατί αν η διαβούλευση είναι μια ανοιχτή διαβούλευση με το κοινό που ξέρει τι θα πει ε, φίνινγκ και είναι κατά του φίνινγκ τότε και πάλι διαπράττουμε ένα σφάλμα γιατί όλοι είμαστε κατά του φίνινγκ αλλά εδώ μιλούμε για την εξαίρεση αυτό είναι το θέμα της συζήτηση. Η κατάργηση αυτής της εξαίρεσης δεν έχει νόημα. Το μοναδικό επιχείρημα που άκουσα και που θα μπορούσε να ευσταθεί κάπως είναι η δυσκολία ελέγχου κατά την εκφόρτωση. Γιατί μερικές φορές, σπάνια βέβαια, αλλά μερικές φορές η εκφόρτωση ε, των ε, πτερυγίων και του κορμού του Καρχαρία, του σώματος του Καρχαρία, δεν γίνεται ταυτόχρονα στο ίδιο λιμάνι, γιατί ε, σε άλλο λιμάνι προορίζονται τα πτερύγια και σε άλλο το υπόλοιπο σώμα του Καρχαρία. Αν όμως το πρόβλημα είναι πρόβλημα ελέγχου, τότε δικό μας έργο είναι να βρούμε μηχανισμούς για να ενισχύσουμε τον έλεγχο και να μην αναζητήσουμε την απλούστερη λύση. Έχουμε πρόβλημα ελέγχου, άρα τα καταργούμε όλα, πονάει δόντι, βγάζουμε δόντι. Αυτή παρά είναι απλοϊκή η λύση. Σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα προβλήματα της αλίας. Γιατί να κατοργήσουμε μία εξαίρεση θίγοντας ένα συγκεκριμένο τμήμα του αλληλευτικού στόλου που ασχολείται με αυτή την αλία. Ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική και διαπιστώνουμε ότι περιορίζουμε όλο και περισσότερο και σφίγγει ο κλειός γύρω από την αλία και με πιο λογικό επιχείρημα θέλουμε να περιορίσουμε ή να καταργήσουμε μια εξαίρεση που είναι και λογική ούτως ή άλλως μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Αν υπάρχει λυπής έλεγχος, να βρούμε μηχανισμούς για να γίνει πιο αποτελεσματικός και αυστηρός. Γιατί η βούληση όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κοινού είναι ε, να καταπολεμήσουμε την πρακτική του φίνινγκ. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Η εξαίρεση άλλο νόημα έχει. Και η κατάργηση εξαίρεσης δεν είναι λογική εδώ. Δεν είναι εύλογη. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ναι και δεν έχουμε και χρόνο, δεν ε, πρόκειται να επισέλθω σε πιο λεπτομεριακή ανάλυση και σε επιχειρήματα υγείας ή κινδύνων ε, κατά των ναυτικών ή σε φυτογειονομικά θέματα, σε θέματα αποδοτικότητας. Θα έχουμε άλλη ευκαιρία και πολύ περισσότερο χρόνο για να επισέλθουμε στα θέματα αυτά, αλλά πιστεύω ότι σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων δεν είναι σκόπιμο να επισέλθουμε σε λεπτομέρειε. Θα ήθελα πάντω να πω στου συναδέλφου ότι δεδομένη τη ευαισθησία αυτού του θέματο ε, ε, γράφω ένα ενδιάμεσο έγγραφο, όχι την έκθεσή μου, ένα ενδιάμεσο έγγραφο εργασία και συζήτησης, ώστε με εμπεριστατωμένο τρόπο με σαφήνεια και χωρίς συγκινησιακή φόρτιση να εγκύψουμε στο θέμα και να δούμε ποιο είναι το διακύβευμα και πώς θα πρέπει να δράσουμε προκειμένου να α, τηρήσουμε αυτή την α, κοινή μας θέση που είναι η καταδίκη αυτής της πρακτικής. Επαναλαμβάνω, η πρώτη ανταλλαγή απόψε, κύριε Πρόεδρε, προβλέπεται για τα τέλη Φεβρουαρίου, μεταξύ 27 και 29 Φεβρουαρίου. Το έγγραφο εργασίας ε, θα υποβληθεί στις 21 Μαρτίου. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στις 24 και 25 Απριλίου. Η διορία για την υποβολή των τροπολογιών ε, λίγη στις 27 Απριλίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα στις 30 Μαΐου. Θα μοιράσω, επαναλαμβάνω, και αυτό το έγγραφο εργασίας, το μεταβατικό κατά κάποιο τρόπο και θα οργανώσω και μία συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές, ώστε με νυφάλιο και ψύχρεμο τρόπο να εξετάσουν αυτό το ζήτημα και ελπίζω ότι θα βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τον έλεγχο, γιατί τελικά αυτό είναι το πρόβλημα, ο ελληπής έλεγχος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμέβα και μετά η κυρία Φράγα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά και την εισηγήτριά μας, την κυρία Πατραονέβες. Ε, προβλέπω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε και τις θέσεις μας. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω και να επιδοκιμάσω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εύστοχη, απαραίτητη και επίγουσα κατά τη γνώμη μου. Γιατί τα στοιχεία που εξετάσαμε τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες το αποδεικνύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις ε, περιοχές που κατεξοχήν ε, εξάγουν φτερή για καρχαρία Προ τι ασιατικέ χώρες και μερικές ε, χώρες, ιδιαίτερα η Ισπανία, είναι συνυπεύθυνε για αυτή την κατάσταση. Είναι, αν όχι αδύνατο, πραγματικά πολύ δύσκολο ο έλεγχος της κατάστασης. Έχουμε μια νομοθεσία που από μόνη της είναι σχετικά όριστη και συγκεχημένη. Το αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν ποσοστά σε όλες σε όλου του τρόπου αλίας και σε όλα τα αλληλευτικά είδη. Δεν ισχύουν ενιαία κριτήρια και το 5% που έχουμε στον κανονισμό μας ούτω ή άλλω είναι το διπλάσιο άλλων χωρών και άλλων ζωνών όπω του Καναδά. Ε, Εκεί το 5% αφορά το, το καθαρό βάρος, ενώ το δικό μας 5% αφορά το συνολικό βάρος. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια λύση θέλουμε μία συζήτηση και σίγουρα α, τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού και νομίζω ότι η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε για να ρυθμίσουμε σωστά αυτή τη πρακτική και αυτά τα αλλιεύματα χωρίς τις ολέθριες συνέπειες του φίνινγκ. Ολοσχερή απαγόρευση, χωρίς καμία εξαίρεση, είναι ο μοναδικός τρόπος για να ε, εφαρμόσουμε την πολυσύνθετη αλλά απαραίτητη αυτή νομοθεσία. Μόνο με ολοσχερή απαγόρευση και χωρίς καμία εξαίρεση μπορούμε να έχουμε και οικονομικά αποτελέσματα, γιατί πραγματικά υπάρχει τεράστια διαφορά οικονομική μεταξύ της αξίας των πτερυγίων και της αξίας του υπόλοιπου σώματος του Καρχαρία. Και η απαγόρευση του διαχωρισμού των πτερυγίων από το σώμα του Καρχαρία είναι πολύ θετική. Γι' αυτή είναι η θέση μας λοιπόν. Είμαστε κατά της εξαίρεσης και άρα υπέρ της κατάργησης. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση και θα δούμε τι μόρφη θα έχει τελικά το έγγραφο εργασίας. Πάντως θα θέλαμε ευθύ εξ αρχής να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτή, αυτή την κατεύθυνση θα έχουν και οι τροπολογίες μας και αυτό το ύφο. Η ε, κυρία Φράγκα, κύριε... ε, ε Ρωμέβα, θα ήθελα να σας πω, η λύση πονάει δόντι, βγάζει δόντι, δεν είναι η κατάλληλη. Δεν μπορούμε, επειδή έχουμε πρόβλημα ελέγχου, να καταργούμε ολόκληρη την πρόταση. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος να γίνει ό,τι μορφή και αν έχει πρόταση. Γιατί χωρίς έλεγχο η κατάσταση θα είναι ακόμη χειρότερη. Νομίζω ότι είναι ε, η πρόταση αυτή ένα καλό παράδειγμα της υποταγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο στι πιέσει από μη κυβερνητικέ οργανώσει, γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και φαίνεται ότι υπέκυψε στι πιέσει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφάσισε να υποβάλει τροποποίηση. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη, την ισχύουσα νομοθεσία, η ισχύουσα νομοθεσία δεν τηρείται. Μα το λένε και οι εμπειρογνώμονε. Και γνωρίζει ο κ. Ρωμέβα ότι ε, η Ούτε η Ισπανία τήρει αυτή την νομοθεσία. Και ένας εμπειρογνώμονας κορυφαίος στο... που έχει εξετάσει την περίπτωση εκατομμυρίων καρχαριών είπε στο ICAT ότι όχι μόνο η αφαίρεση των πτερυγίων, αλλά μερικές φορές και το είδος του καρχαρία επηρεάζει ε, την αναλογία της αξίας μεταξύ πτερυγίου και σώματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλιεύονται μόνο δύο είδη καρχαρία. Οπότε για μας το θέμα είναι πολύ πιο απλό. 80% είναι ένα είδο καρχαρία και 20% άλλο είδο καρχαρία. Και μάλιστα τα παραγαδιάρικα πλοία αλλιεύουν αυτά τα δύο είδη καρχαρία. Και στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό ε, πρόκειται για αλληλευτικά είδη που δεν απειλούνται από εξαφάνιση και η βιομάζα τους είναι σε υψηλό επίπεδο. Άλλωστε, ούτε από βιολογική άποψη είναι αλληλευτικά ηχθή από θέματα που διατρέχουν κίνδυνο. Άλλωστε, δεν χάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα παραγαδιάρικα που αλλιεύουν αυτές, αυτά τα, τα είδη είναι λίγα. Άλλωστε στην Ισπανία καταναλώναμε καρχαρία πολύ πριν θεσπιστεί η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ρωμέβα γνωρίζει την αλήθεια. Ε, στην Ισπανία και Πορτογαλία καταναλώναμε καρχαρία χρόνια ολόκληρα. Και εξάγουμε και σε άλλες χώρες, γιατί και άλλες χώρες το καταναλώνουν. Δεν είναι θέμα μόνο πτερυγίων, αλλά θέμα και σώματος, του υπόλοιπου σώματος του κορμού του καρχαρία η ευρωπαϊκή βιομηχανία, η ευρωπαϊκή ελίδα e δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το φίνινγκ. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν πρόβλημα με το φίνινγκ. Αλλά αν έχουν πρόβλημα να στραφούν προς ασιατικέ χώρες. Αυτές είναι που κάνουν φίνινγκ, όχι οι ευρωπαϊκές. Η Επίτροπος είπε ότι χάρη στην κοινοτική νομοθεσία ε, καταργήθηκε η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει την άγνοια τη. Ε, Επιτρόπου Αλία για τι πρακτικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η φίνιγκ ούτω ή άλλω δεν γινόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν την νομοθεσία. Δεν ξέρω πώ θα λύσουμε το πρόβλημα. Πάντω, εγώ διάβασα τη μελέτη επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι η τελευταία πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, καταστροφική για, τα, για το στόλο παραγαδιάρικων. Κύριε Ρωμέβα, και το κόστος θα είναι τεράστιο. Σας παραπέμπω στη, στα στοιχεία και δημιουργεί και μια σειρά προβλημάτων. Τώρα, η μερική κοπή των πτερυγίων ε, και η συνέχιση, η ολοκλήρωση ε, της κοπής στη γη, αυτό, αυτό επιδεινώνει την κατάσταση ε, του προϊόντος στο τέλος και, και φθήνει το προϊόν. Άρα η ποιότητα υποβαθμίζεται και άρα και η τιμή του προϊόντος θα μειωθεί. Και υπάρχει και το θέμα της αλυσίδας του ψύχους. Γιατί σε πολλά από τα λιμάνια της εκφόρτωσης, στο πράσινο ακροτήριο για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ψυκτικές εγκαταστάσεις για να ε, μην διακοπεί η αλυσίδα του ψύχους. Οπότε, αν διακοπεί ε, η αλυσίδα του ψύχους, χαιρετίσματα για την ποιότητα του προϊόντος. Τώρα μπορούμε να έχουμε κατάλογο των χωρών εκφόρτωση. Βλέπετε ότι οι περισσότερε χώρε δεν έχουν τέτοιε εγκαταστάσει ε, που να εξασφαλίζουν την ψήξη. Επίσης, ε, ε, λέμε η μεταποίηση στη γη των προϊόντων ε, να υπάγεται στην υποχρέωση πιστοποίηση από τις αρχές της χώρας εκφόρτωσης. Στις χώρες αυτές όμως είναι πολύ δύσκολο να λυθεί τέτοια πιστοποίηση. μετά, η οριστικός διαχωρισμός των πτερυγίων από το σώμα του καρχαρία στη γη που έχει ξεκινήσει το σκάφος, κάτι τέτοιο προϋποθέτει αλλαγή και της προέλευσης του προϊόντος. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Μία σειρά προβλημάτων δημιουργεί η πρόταση. Θα πρέπει να τα αναλύσουμε όλα αυτά για να δούμε ποια είναι η κατάλληλη λύση. Και για να μην πλήξουμε τον αλληλευτικό μας κλάδο. Επαναλαμβάνω, η λύση πονάει εδώ το βγάζουμε, δεν είναι η κατάλληλη λύση. Δεν μπορούμε να αποδεκατήσουμε τον κλάδο μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο. Απλώς να πετήσουμε αποτελεσματική νομοθεσία και σωστή εφαρμογή της. Χωρί να πλήττει ένα τομέα, το τομέα των παραγαδιάρικων, που ούτως ή άλλως είναι πολύ επιλεκτικός. Και με τα δύο είδη καρχαρία πολιεύονται δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε βιωσιμότητα ούτε βιοπικιλότητα. Επαναλαμβάνω, κύριε Ρωμέβα, είστε λογικός άνθρωπος, είστε και σκιωδησηγητή. Θα το συζητήσουμε με ψύχρεμο και λιφάλιο τρόπο για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Θεοφίλου, θέλετε να επανέλθετε. Ή ο κύριος Ντέβι, συγγνώμη, δεν σας είχα δει προηγουμένως. Κύριε Ντέβις, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περιγράφει ως ε, ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εμένα μου φαίνεται πολύ οικία. Την είχαμε πριν 8 χρόνια όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός αυτός. Ε, θυμάμαι ότι τότε διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσει όπω η Shark Trust έλεγε ότι πρέπει να εκφορτώνει κανεί ε, τον Καρχαρία ολόκληρο για να μπορεί να ελέγχει τα νούμερα. Ε, και Εκείνη την εποχή η Κομισιόν είχε πει όχι και ε, προέβαλε πολλά από τα επιχειρήματα τα οποία μόλις ε, αναφέρθηκαν. Αλλά τώρα η Κομισιόν επανέρχεται και λέει «Κάναμε λάθος. Κάναμε λάθος τότε. Πρέπει να διορθώσουμε το λάθος μας. Πρέπει να εκφορτώνουμε τους καρχαρίες ολόκληρους. Δεν λειτουργεί το σύστημα και ξέρουμε γιατί δεν λειτουργεί. Διότι ο κόσμος εξαπατά, λέει ψέματα. Ε, και δεν θα πρέπει να χρειάζεται να ε, δαπανούμε περισσότερα χρήματα για τους ελέγχους. Πάντα ήταν δύσκολο το θέμα αυτό, γι' αυτό ακριβώς το επιχείρημα ήταν να εκφορτώνουμε ολόκληρο τον Καρχαρία. Ε, η κυρία Φράγα είπε ότι οι καρχαρίες δεν τα περνάνε και πολύ άσχημα ως είδος, δεν απειλούνται. Δύο είδη καρχαριών. Εγώ έχω αμφιβολίες χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν συνάντησα καρχαρία πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ε, ε, πολλαπλασιάζονται πολύ αργά και η έκθεση λέει, της Κομισιόν λέει ότι οι καρχαρίες απειλούνται ε, ως ε, αποτέλεσμα της αυξημένης ε, ζήτησης προϊόντων καρχαρία, ιδιαίτερα των πτερυγίων. Ελπίζω η Κομισιόν να μ' ακούει, διότι πρέπει τα στοιχεία να βασίζονται στην επιστήμη. Προσωπικά, θα βάλω το πράσινο καπέλο μου εγώ πολύ ευχαρίστω ε, θα ήθελα να δω απαγόρευση τη ε, πώληση περιγείων καρχαρία. Ε, αλλά να κάνουμε τουλάχιστον αυτό το μετριοπαθέ βήμα. Ο κύριο Θεοφίλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να μπω σε ε, αναλυτική συζήτηση σχετικά με τα επιστημονικά επιχειρήματα στη συζήτηση αυτή. Σύντομα θέλω να σας αναφέρω ότι τα δεδομένα που υπάρχουν για τα δύο βασικά είδη που ε, αλλιεύουν ε, τα, τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι πολύ καλής ποιότητας, δεν έχουμε πολύ καλά στοιχεία, πολύ σαφή στοιχεία και αναγνωρίζουμε ότι το καθεστώς των δύο αυτών ειδών ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Υπάρχουν κάποια αποθέματα ε, υπάρχουν διάφορα αποθέματα με, σε διαφορετική κατάσταση. Ε, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα πιο συγκεκριμένα θέματα που ε, ανέφεραν οι τέσσερις βουλευτές που πήραν το λόγο. Καταρχήν, ο κανόνας ε, που έχουμε για το 5% ε, αντικατοπτρίζει τον κανόνα 5% που έχουν οι ICAT και οι IOTC που είναι οι οργανισμοί που ελέγχουν ε, τις περιοχές όπου πολλά από τα ισπανικά και πορτογαλικά παραγαδιάρικα ψαρεύουν. Αναφέρεται, αναφέρει λοιπόν ο κανόνας ότι το ε, βάρος των πτεργείων δεν ε, πρέπει να ξεπερνάει το 5% του αλιεύματος χωρίς να ξεκαθαρίζει αν ε, μιλάμε για το, ε, το, το βάρος ζωντανών ψαριών. Εμείς αυτό επιλέξαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπει δηλαδή τα, στα σκάφη να διατηρούν πάνω στο σκάφος δύο ή τρία δύο-τρεις φορές το βάρος ε, που θα επιτρεπόταν αν, συγκρίναμε, αν χρησιμοποιούσαμε ως μέτρο το το βάρο των ψαριών αφού έχει κοπεί το κεφάλι και διάφορα άλλα μέρη του. Είχαμε λοιπόν στο παρελθόν κάποια προβλήματα με τον κανόνα αυτό, διότι άλλα κράτη-μέλη της ICAT και της IOTC ε, εφήρμοσαν αυτόν τον διαφορετικό κανόνα ε, των ειδικομένων ψαριών, καθαρισμένων ψαριών. Οπότε... Ε, κλήθηκε η Κομισιόν να παρέμβει υπέρ αυτών των Ισπανικών ε, και Πορτογαλικών πιθανότατα σκαφών, στον Τέρμπαν και αλλού δεν θυμάμαι. Ε, σίγουρα θυμάμαι ότι ε, πρόκειτο για κάποια Ισπανικά σκάφη. Κλήθηκε λοιπόν η Κομισιόν να παρέμβει υπέρ των σκαφών αυτών που ξεπέρασαν το βάρος στα λιμάνια εκφόρτωσης. Αν καταργήσουμε λοιπόν ε, το, την αναλογία αυτή του 5% λύνουμε το πρόβλημα για τον ε, στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον από το 2009 και μετά μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία συνεχίζουν ε, να εκδίδουν ειδικέ άδειε αλληλείας. Άλλα κράτη-μέλη που στο παρελθόν εξέδιδαν τέτοιες ε, τέτοιες άδειες ε, σταμάτησαν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Λιθουανία. Προφανώς λοιπόν αυτά τα κράτη-μέλη βρήκαν τρόπο να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν από εκφορτώσεις σε λιμάνια τρίτων χωρών χωρίς να έχουν όλες τις, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ε, επιπλέον την προηγούμενη εβδομάδα το Ταϊβάν που είναι μία από τις χώρες που ε, συχνά ε, κατηγορούμε για το φίνινγκ και, και το σκότωμα καρχαριών ε, ε, ε, εξέδωσε έναν κανονισμό για την ε, εκφόρτωση του συνόλου του καρχαρία χωρίς να έχει καμία επεξεργασία. Άλλες χώρες, η Κωνσταντίνα, η Αυστραλία είχαν εδώ και χρόνια πολιτική να εκφορτώνεται το ψάρι μαζί με το πτερίγιο και άλλες χώρες έχουν συζητήσει τη δυνατότητα αυτή στην ICAT και στην IOTC. Υπάρχει Υπάρχει λοιπόν μια γενική τάση, δεν αποτελεί μόνο έκκληση μη κυβερνητικών οργανώσεων, αποτελεί γενική τάση ε, στις ε, διάφορες περιφερειακές ε, οργανώσεις διαχείρισης της αλληλείας για εκφόρτωση του καρχαρία με το πτερίγιο. Εάν λοιπόν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θα είμαστε σε θέση να στηρίξουμε και άλλες χώρες σε διεθνή φόρουμ ε, για να ακολουθήσουν και εκείνη αυτή την κατεύθυνση. Ε, Κυρία Πατράου, εγώ έθεσα μια συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μου απάντησε όμως. Ακούσαμε ότι η πρόταση ε, ήταν ο καρπός μιας δημόσιας διαβούλευσης. Ρώτησα λοιπόν, ποιος συμμετείχε στη διαβούλευση αυτή και ήταν ενήμεροι όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση, γιατί όλοι είμαστε κατά του φίνινγκ. Αυτή όμως η δημόσια διαβούλευση, ίσως ε, ήταν ε, εμπειρογνώμονες, ίσως απλώς ε, ήταν κατά του φίνινγκ, γι' αυτό τάχθηκαν και υπέρ της κατάργησης της αφαίρεσης. Ρώτησα λοιπόν ποιοι ακριβώς συμμετείχαν στη διαβούλευση. Όπως είπα και στην αρχή στους συναδέλφους, δεν ε, ασχολήθηκα με το περιεχόμενο, με την ουσία. Αυτή, το θέμα επίγει, είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν χρειάζεται στην πρώτη ανταλλαγή να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Είπα ότι θα ήθελα νυφάλια και ψύχρεμα να συζητήσουμε το έγγραφο που θα υποβάλω αργότερα, γιατί φάνηκε ότι ο κόσμος δεν, ξέρει, δεν γνωρίζει με ακρίβεια τα επιστημονικά πορίσματα για το θέμα αυτό. Εμείς έχουμε ευθύνε. Και μία από τις ευθύνες μας υποθέτει ε, η λήψη, η θέσεων και η λήψη αποφάσεων εμπεριστατωμένα όμως, με γνώση της κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τα επιστημονικά στοιχεία, να γίνουν πολλές συνεδριάσεις, να υποβληθεί ένα πρωτόλιο εργασία, να ακούσουμε τα επιχειρήματα των ΜΕΝ και των ΔΕ και να επιδιώξουμε μια συνενετική λύση στην Επιτροπή μας. Φυσικά θέλουμε βελτίωση του ελέγχου. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτό που είπατε ότι δεν θέλουμε να δαπανίσουμε χρήματα για έλεγχο. Γιατί αν είχαμε ένα κανόνα για όλα τα, ένα κανόνα για όλα τα σκάφη, μόνο να κάναμε οικονομίες στον έλεγχο. Ο έλεγχος μας ενδιαφέρει. Μην μου λέτε λοιπόν θέλω να δαπανίσω κονδύλια για τον έλεγχο, επειδή πρόκειται απλώς για πτερή, για καρχαρία και δεν ε, εμπλέκονται εδώ όλα τα ελευτικά σκάφη, τότε θα ήταν πολύ πιο γενναιόδοροι στον έλεγχο. Επαναλαμβάνω, να επενδύσουμε σε συστήματα ελέγχου, ώστε να μην υπάρχουν διαρροές, ε, να μην υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και επιπλέον Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006 είχαμε δηλώσει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζεται το φίνινγκ, δεν εφαρμόζεται αυτή η πρακτική. Οπότε προσοχή, από τη μια μας λέτε ότι δεν γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το φίνινγκ και από την άλλη λέτε μπορεί να γίνεται αλλά δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Θέλουμε εμπεριστατωμένε ε, μελέτες ε, και επιστημονικά πορίσματα για να διαμορφώσουμε τη γνώμη μας. Ευχαριστώ κύριε Πατράου. Θα συνεχίσουμε τόσο άλλους τη συζήτηση για το θέμα αυτό και θα μπορέσει τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει πιο λεπτομεριακά. Για τα διάφορα δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο. 28. Ανακοινώσει του Πρόεδρου σχετικά με τι αποφάσει που έλαβαν οι συντονιστέ. Έχετε λάβει, αν δεν κάνω λάθο, τι αποφάσει των συντονιστών. Οπότε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, παρακαλώ να εγκρίνουμε τι αποφάσει των συντονιστών. Επόμενη συνεδρίαση 27, 28 και 29 Φεβρουαρίου. Αυτά. Ευχαριστώ θερμά όλους ε, τους συμμετέχοντες στη συζήτηση και τους διερμήνεις. Ε, ήσταν πολύ ευγενικοί γιατί ήταν και η παρθενική μου προεδρία σε αυτή την ε, πολύ ωραία συνεδρίαση. Ευχαριστώ. για τη συνεδρίαση. Καλό σας μεσημέρι.